Bene. Ε, eh, e eh. Κυρίε και κύριοι, θα μιλήσω Ιταλικά, οπότε παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. Να κηρύξουμε την έναρξη της ακρόασης αυτής της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτών. Και να καλωσορίσω τον υποψήφιο επίτροπο την Ναύρατσιτ να κάνω κάποιες αναρκτήριες παρατηρήσεις, διότι η ακρόαση αυτή, όπως τα ξέρει και εκείνο, είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική. Όχι μόνο όμως για την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, αλλά και για την παρουσία των συναδέλφων από τις Επιτροπές Ήτρε και την Επιτροπή ΠΕΤΗ. Η είναι επιτροπή που θα συμμετάσχει, ενώ η Επιτροπή ΠΕΤΗ είναι απλώς παρατηρήτρια. Αυτός ο συνολικός, ο ομαδικός χαρακτήρας της ακροασής μας δείχνει ότι ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα έχουν αξία αυταπόδεικτη ως αυτούσιες αρχές, αλλά και οικονομικές προεκτάσεις, καθώς και κοινωνικές. Έτσι λοιπόν οι εκπαιδευτικές πολιτικές και οι πολιτικές μάθησης έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες που θα προσφέρουμε στους νέους. Το ίδιο και για την πολιτική για τους νέους που είναι κεντρική σημασία για τη στρατηγική 2020. Αυτό σημαίνει ότι για μας τα θέματα αυτά είναι ζωτική σημασία για την υλοποίηση των αρχών της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για να κατανοήσουμε ποιο είναι το όραμα της Ευρώπης που έχουμε σήμερα και ποιο ανθρώπινο, πολιτικό και κοινωνικό κεφάλαιο προτείνουμε στους πολίτες σήμερα. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Ναύρατσιτς, δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι ανησυχίες, οι εκκλήσεις που μας έχουν απευθυνθεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά και αυτούς τους μήνες, από πολλούς πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών. Σήμερα θα έχετε κάθε ευκαιρία, και θα το φροντίσουμε εμείς αυτό, σε αυτήν την ακρόαση να υπάρχει ο μέγιστος δυνατός αμοιβαίος σεβασμός. Θα έχετε λοιπόν κάθε ευκαιρία και το εύχομαι να μας καθησυχάσετε για το ότι και εσείς ε, ε, σέβεστε απολύτως τις αρχές της συνθήκης και ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές μας θα ε, χαραχθούν μέσα στην πλήρη ανεξαρτησία την προσωπική σας και στο ρόλο σας ως Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω τη διαδικασία προβλέπεται σήμερα για την διεξαγωγή αυτή τη ακρόαση. Όπω τα γνωρίζετε, οι κατευθυντήρε γραμμέ για τι ακροάσει των υποψήφιων επιτρόπων περιλαμβάνονται στο παράδειγμα 16 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου, όπου λέγεται το εξή. Το Κοινοβούλιο αξιολογεί του υποψηφίου επιτρόπου βάσει των γενικών του ικανοτήτων, τη ευρωπαϊκή του δέσμευση και τη προσωπική του ανεξαρτησία αποτιμά τη γνώση του μελλοντικού χαρτοφυλακίου που θα αναλάβουν και τις δυνατότητες επικοινωνίας τους. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για την ακρόασή μας. Ε, σας ευχαριστώ κύριε υποψήφια Επίτροπε που ήδη απαντήσατε σε κάποιες προκαταρκτικές ερωτήσεις που σας απεστάλησαν. Οι απαντήσεις σας έχουν διανεμηθεί σε όλα τα μέλη, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Και συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο με τα έγγραφα για τη σημερινή ακρόαση μαζί με το βιογραφικό σας. Σε αυτό το σημείο θα έλεγα να οργανώσουμε τη συζήτηση ως εξής. Αρχικά, ο υποψήφιος επίτροπος Ναύρατσιτ θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει 15 λεπτά για τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε, θα έχει θα υπάρξει χρόνος για 45 ερωτήσεις από τους ε, συναδέλφους βουλευτές και η συζήτηση θα βασιστεί στην αρχή ping-pong όπως ονομάστηκε, δηλαδή παρεμβάσεις τριών λεπτών συνολικά η κάθε μια. Ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση του Επιτρόπου σε κάθε ερώτηση. Να θυμίσω ότι ο πρώτος γύρος ερωτήσεων θα τεθεί από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και από τους μη εγγεγραμμένους. Και ε, θα ακολουθήσει η Επιτροπή η η οποία συμμετέχει στην ακρόαση αυτή, ενώ η Επιτροπή Αναφορών ΠΕΤΗ είναι απλώς προσκεκλημένη. Μόλις ολοκληρωθεί ο γύρος ερωταπαντήσεων, στο τέλος ο υποψήφιος επίτροπος θα έχει πέντε λεπτά στη διάθεσή του για μια καταληκτήρια παρέμβαση και οι γλώσσες που θα καλυφθούν σήμερα από, την από τη Διερμηνία είναι 23. Μπορούν οι ομιλητές να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα τους εκτός από τα μαλτέζικα. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους. Η ακρόαση θα μεταδοθεί απευθείας στο διαδίκτυο του Κοινοβουλίου και επίσης εκεί θα υπάρχει και βιντεοσκοπημένη η ακρόαση. Επειδή θα μεταφράζεστε ταυτοχρόνως από τους διερμηνείς, παρακαλώ να μιλάτε με έναν φυσιολογικό ρυθμό. Να καλωσορίσω λοιπόν και πάλι τον κύριο Ναύρατσιτς και του δίνω το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ.